Bien. Bonjour. Καλή σας μέρα. Ελπίζω να είστε σε φόρμα σήμερα το πρωί. Αρχίζουμε εκ νέου τις εργασίες μας εκεί όπου σταματήσαμε χθες. Σήμερα το πρωί θα εξετάσουμε τη γνωμοδότηση του κ. Ντόρφμαν τον οποίο χαιρετίζω για τις μεταβατικές διατάξεις ε, για τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη του ΦΕΑ του ΦΕΑΝΤΕΡ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργίας ε, Εγγυήσεων του ΦΕΑΓΑ ε, για το 2021. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020 είναι ακόμα από διαπραγμάτευση. Είναι λοιπόν απαραίτητο για να εγγυηθούμε μια ομαλή μετάβαση να εγκρίνουμε μεταβατικά μέτρα που θα μας επιτρέψουν να επιμηκύνουμε την, την εφαρμογή των υπάρχων κανονισμών έως την ε, θέσπιση του νέου συστήματος. Η υπάρχουσα λοιπόν νομοθεσία πρέπει να τροποποιηθεί για να συμπεριληφθούν μεταξύ άλλων τα ποσά και οι οροφές που θα ισχύσουν ε, και που πρέπει να καθοριστούν για, την, για το επόμενο ΠΔΠ 2021-2027. Ο κ. Ντόρφμαν επαναφέρει τους πόρους για τη γεωργία σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου για την Δελταφή και δημιουργεί επίσης κάποιες διατάξεις ε, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν κάποιες δεσμεύσεις που έχουμε ήδη αναλάβει ε, και για τις οποίες βεβαίως υπάρχουν τα υπάρχοντα κονδύλια έχουν ήδη εξαντληθεί. Θα δώσω λοιπόν ευθύ αμέσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή και μετά στον σκιώδη εισηγητή και βεβαίως μετά θα μιλήσουν και όποια μέλη το επιθυμούν. Κύριε Ντόρφμαν, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται πράγματι για έναν κανονισμό που θα ρυθμίσει την κοινή γεωργική πολιτική για το επόμενο έτος γιατί δεν θα υπάρχει ακόμα του χρόνου η νέα μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ. Οπότε κάνουμε μια γνωμοδότηση προς την ε, Επιτροπή Γεωργίας που είναι η αρμόδια. Είναι τεχνικός κανονισμός για να εγγυηθούμε λίγο πολύ τη συνέχεια της σημερινής πολιτικής και για το επόμενο έτος. Γι' αυτό έκανα ε, λίγες ε, τροπολογίες ε, στην έκθεσή μου γιατί δεν έχει και πάρα πολύ νόημα αφού θα γίνει η γενική μεταρρύθμιση. Γι' αυτό οι τροπολογίες μου επικεντρώνονται κυρίως στα θέματα που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή στον δεύτερο πυλώνα στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης προσπάθησα να κάνω όσο το δυνατόν πιο ευελικτό τον τρόπο εργασίας των περιφερειών να αυξηθεί ο χρόνος λήψη αποφάσεων από 10 στις 30 ημέρες μετά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες τους. Και βεβαίως να δούμε και το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο. Για να δούμε εάν θα τραβήξουμε λεφτά από τον νέο προϋπολογισμό ή τον παλαιό. Κάτι άλλο, η εσωτερική σύγκληση των πληρωμών στον πρώτο πυλώνο πρέπει να συνεχιστεί, όχι μπορεί να συνεχιστεί, είναι υποχρεωτικό δηλαδή και όσον αφορά τη χρηματοδότηση των υπερπόντιων περιοχών και των εξόχως περιφερειακών Γνωρίζω ότι είναι μια επιθυμία βεβαίω, αλλά πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο έχει λάβει ήδη την απόφασή του όσον αφορά τα κονδύλια και πρέπει να το επαναλάβουμε και εδώ. Αυτά με δύο λόγια. Merci beaucoup, monsieur le, le ευχαριστώ κύριε Σίγητα. Έχετε δίκιο. Όντως ε, πρέπει να ασχοληθούμε με τα ζητήματα που αφορούν τη δική μας Επιτροπή και το θέμα της ανάπτυξης υπαίθρου είναι εξαιρετικά σημαντικό ε, μέσα στην γενική ε, συνέπεια και ροή της πολιτικής συνοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ασχοληθήκατε με το θέμα του Ταμείου Ποζέη, γιατί ακριβώς το Ευρωκοινοβούλιο είχε υιοθετήσει στην Ολομέλειά του τη θέση για τη διατήρηση ε, αυτού του Ταμείου. Ε, τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, ε, στους κοιόδες με συγχωρείτε, Ποιο θα ήθελε να πάρει το λόγο, ο κύριο Βερμπίστε. Ευχαριστώ. Η Ιζαμπέλ ε, ε, λυπάται που δεν μπορεί να είναι εδώ, αλλά μου ζήτησε να σας διαβιβάσω τα σχόλιά της. Ο μεταβατικός κανονισμός είναι πολύ αποφασιστική σημασία σε όργανο για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα στη στήριξη του γεωργικού τομέα. Θα διευκολύνει τους γεωργού να συνεχίσουν να σχεδιάζουν τις δραστηριότητε τους. Ε, ταχεία πρόοδο στι διαπραγματεύσει για τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική καθώ και η παράδοση των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών εν θα είναι, πρέπει να παραμένουν προτεραιότητα. Όμω, δεδομένου του σημείου των διαπραγματεύσεων, πιστεύω πω ε, μία σόφρον προσέγγιση σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε προβλεψιμότητα και σταθερότητα για τον τομέα. Ε, από αυτό το φως θεωρώ επίσης ότι η πρόταση που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με, δια της Προέδρου του για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι απογοητευτική και δεν καλύπτει τις προκλήσεις ε, στις οποίες πρέπει να απαντήσει η κοινή γεωργική πολιτική. Συμφωνώ με τον εισηγητή Ντόρφμαν ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς και να αρνηθούμε οποιασδήποτε περικοπές στις, ε, στην περικοδότηση του ΠΟΣΕΙ για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό το πρόγραμμα που είναι ένα ασήμαντο βάρος στο σύνολο του προπολογισμού για τις περιοχές οι οποίες ε, ε, είναι ιδιαίτερα μειονεκτούσες λόγω της γεωγραφικής τους ε, θέσης και λόγω αξεπέραστων διαδομικών ε, περιορισμών ε, και ιδιαιτεροτήτων είναι πολύ σημαντική. σημαντικό το κονδύλι. Επίσης αναγνωρίζεται από τη συνθήκη λειτουργίας του, συγγνώμη, δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η ιδιαιτερότητα. Από το Renew Στεφάν Μπιζού. Καλημέρα σας, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο όνομα της ομάδας Ρινιού θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του και να πω ότι συμμερίζομαι τη δική του άποψη για ανάγκη ευελιξίας στη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Έχετε δει και που επιμένετε και είναι εξαιρετικά σημαντικό να πούμε ότι ε, συμμεριζόμαστε τη δική σας φιλοδοξία απέναντι στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και ειδικά τις υπερπεριφερειακές. Η ιδιαίτερη φύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε γνωρί, μας κάνει να γνωρίζουμε πως χρειάζεται μια ιδιαίτερη ε, παρακολούθηση είναι το νόημα αυτό του άρθρου 349 της συνθήκης. Πρέπει να είμαστε στο ύψος αυτής της φιλοδοξίας της συνοχής, της Ευρώπης, της συνοχής και της αλληλεγγύης. Το να διατηρήσουμε λοιπόν το σημερινό επίπεδο στο, για το ΠΟΖΕΙ είναι μη, μη διαπραγματεύσιμο. Ο πρώην Επίτροπος στη Γεωργία είχε εκφράσει τη στήριξή του για τη διατήρηση αυτού του κονδυλίου ε, και στη γνωμοδότηση ο εισηγητής προτείνει να επανέλθουμε στο σημερινό επίπεδο του προπολογισμού. Θα καταθέσω δύο ακόμα ε, τροπολογίες. Το πρώτο για να αντισταθμιστεί το κόστος που συνδύεται με το ε, ε, απομακρυσμένη γεωγραφικά θέση όσον αφορά τον έναν υφοδιασμό και έπειτα για να δούμε τη δομή των διαφόρων ε, τομέων στις απομακρυσμένες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να επαγρυπνούμε για τα μεταβατικά αυτά μέτρα της κοινή γεωργικής πολιτικής και φυσικά όλα αυτά αφορούν απασχόληση, περιβάλλον, αλλά ο αγώνας που θα πρέπει να μας ενώσει είναι ο αγώνας υπέρ της ποιότητας των τροφίμων και η ποιότητα ζωής που θέλουμε για μας και για τα παιδιά μας. Δηλαδή είναι ένα θέμα επιβίωσης και γι' αυτό ε, ακριβώς Όλοι ε, πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό το κοινό στόχο. Τελευταία παρατήρηση αφορά τις φιλανδικές περιφέρειες. Νομίζω πως ε, θα πρέπει να επιτραπεί η έγκριση των επιδοτήσεων στη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Ευχαριστώ πολύ, Στεφάν. Εξ ονόματος του, των Πρασίνων, ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα για τις περιφέρειες και πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης αλλά και τις άμεσες ενισχύσεις που σχετίζεται με την ε, δυνατότητα των περιφερειών να επιζήσουν. Έχει μεγάλη σημασία η ευρωπαϊκή βοήθεια για εισόδημα, για ανάπτυξη και βεβαίω η βοήθεια δεν θα πρέπει να μειωθεί. Θα πρέπει να υπάρχει στήριξη του Κοινοβουλίου σε αυτό. Όταν υπάρχει αδυναμία των κρατών να συνεισφέρουν σε νέα προγράμματα. Είμαι σκιώδης εισηγητής ε, στην Επιτροπή Γεωργίας και θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε προβλήματα άμεσων πληρωμών στους αγρότες πρέπει να έχουν ευελιξία εάν δεν, δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε ε, για την ΚΑΠ ε, σε ένα έτος πρέπει να εφαρμόσουμε αυτομάτως παράταση του προηγούμενου έτους. Οι εισηγητές ανέφεραν την ανάγκη να συνεχιστεί η σύγκληση όχι μόνο εσωτερική αλλά και εξωτερική στην περίοδο 2014 έως 2020 υπάρχει μια σύγκληση και θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνει μέχρι το 2027. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά ήμουν εισηγητής για τα στρατηγικά σχέδια και χαίρομαι για το ότι είχε υποστηριχθεί η πρότασή μου και ελπίζω η Επιτροπή αυτή σε αυτήν την θητεία να λάβει υπόψη τις αποφάσεις ε, που ελήφθησαν στο προηγούμενο κοινοβούλιο. Οι κοινότητες επίσης ε, της υπαίθρου πρέπει να εμπλακούν πιο ενεργά. Η νέα ε, ΚΑΠ βεβαίως βάζει τα θεμέλια. Η τρέχουσα όμως όχι. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για την συμπερίληψη, ένταξη των κοινοτήτων της υπαίθρου. Η ευελιξία επίσης πρέπει να προβλεφθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ότι τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία έχουν εξαντλήσει τα κονδύλια πρέπει να εφαρμόσουν όλα τα προγράμματα σε ένα έτος. Αυτό δεν είναι εφικτό στην πράξη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν επιλογή να εστιάσουν μόνο στα προγράμματα προτεραιότητας και να τα εφαρμόσουν πλήρως. Σημαντική επίσης η οικολογική γεωργία και η πρόταση να επεκταθεί ο προγραμματισμός στα τρία χρόνια της Κομισιόν είναι απαράδεκτη. Αλλιώς το 2029 θα σταματήσει. πρέπει λοιπόν να έχουμε του ίδιου κανόνε που έχουμε τώρα και αυτέ τι προτάσει θέλουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ και την ομάδα ID Ιζαμπέλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω Ιταλικά. Μια σύντομη τεχνική σημείωση, άμα επιτρέπετε, μετά από το Brexit Η τέταρτη ομάδα είναι η ID όσον αφορά τη σύνθεση και τον αριθμό των πολιτικών ομάδων. Οπότε πιστεύω θα πρέπει να λάβετε υπόψη αυτή τη διαφορετική σειρά. Σας παρακαλώ λοιπόν να το λάβετε υπόψη στη συνέχεια. Ε, τούτου λεχθέντους επί της ουσίας της πρότασης η ομάδα ID ε, στηρίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός μεταβατικού κανονισμού. Θεωρώ επίσης πως... Το σημείωμα των σοσιαλιστών δημοκρατών για παράταση κατά δύο έτη είναι κάτι το οποίο στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε δεδομένης της αβεβαιότητας ε, των χρονικών ε, ε, πλαισίων εντός των οποίων θα καταφέρουμε να οριστικοποιήσουμε την νέα κοινή γεωρική πολιτική. Έπειτα, συμφωνώ με τα ιστροπολογίες του, του εισηγητού Ντόρφμαν που θέλει να καταστήσει πιο ευέλικτη και αυτή την, ε, αυτές τις διατάξεις ώστε να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια η νομοθετική και καλύτερη προστασία της Ευρωπαϊκής ε, Γεωργίας. Είναι κάτι, είναι ένα στοιχείο που υποστηρίζει η ομάδα μας απολύτως. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με τις τροπολογίες που είδα, ειδικά την τρία που προβλέπει την εκχώρηση κονδυλίων σε περιπτώσεις κρίσης και κατά τα λοιπά επιφυλασσόμεθα να εισάγουμε, να καταθέσουμε περαιτέρω τροπολογίες βέβαια στο βαθμό του δυνατού δεδομένης της φύσης αυτού του κανονισμού ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το χώρο και να εντάξουμε ίσως κάποια περαιτέρω προσθήκη ώστε να βελτιώσουμε και να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Έχετε... Ευχαριστώ. δίκιο. Θα ζήσω από τη γραμματεία να ακολουθεί τη σωστή σειρά. Να θυμίσω πάντως ότι η ομάδα ID δεν μας έχει πει ποιος είναι ο σκιώδης εισηγητής για αυτή την έκθεση. Αν είστε εσείς, εμείς θα το σημειώσουμε αυτό βεβαίως. Ναι, νομίζω ότι στείλαμε ένα mail χθες θα το επαληθεύσω. Πολύ ωραία. Μάλιστα, εσεί είστε λοιπόν σκιώδη συγκήτρια για αυτή την έκθεση. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Μαρτίνα Μίτσελ ε, για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ τον συγητή και με στηρίζουμε τη μεταβατική διάταξη. Θα ήθελα όμω να πω κάτι Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι το φοβερό αυτό το οποίο κάνουμε. Αυτές οι μεταβατικές ρυθμίσεις είναι αποτέλεσμα ότι δεν έχει ακόμα αλλάξει το σύστημα Ευρωπαϊκή Ένωση και τα έχουμε συζητήσει αυτά στην Επιτροπή μας. γι' αυτό χρειάζονται αυτές οι μεταβατικές ε, ρυθμίσεις. Είναι λοιπόν ένα πρώτο αναγκαίο βήμα, αυτό το οποίο στηρίζουμε, για να σώσουμε ε, ό,τι μπορεί να σωθεί, ας πούμε. Ευχαριστώ για αυτή την ε, απαραίτητη υπενθύμηση. Ο συνάδελφος Κρίστοφ Γιώργελ έχει στήσει το λόγο. Του δίνω το λόγο ευθύ αμέσως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κάποια από τα σχόλια που ήθελα να υποβάλω για αυτή την πρόταση είναι τα εξής ε, για τις μεταβατικές αυτές διατάξεις. Οι μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με δαπάνες της προηγούμενης πραγματικής περίοδου, άρθρο 6 του σχεδίου, νομίζω ότι είναι πολύ περιοριστικές, πολύ περιορισμένες μάλλον, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στην ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν, να συνεχίσουν οι πληρωμές με βάση τις απαιτήσει που προκύπτουν από τον οριζόντιο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την μεταρρύθμιση κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Σημαίνει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να επαναπρογραμματίσουμε κάποιες δράσεις για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια συνέπεια με τη νέα πρόταση, μετά τη μεταρρύθμιση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερο διοικητικό άχθος. Και βεβαίως θα έχουμε και αλλαγές ότι αφορά τους δικαιούχους και ότι θα λαμβάνουν η πολωνική κυβέρνηση θεωρεί ότι όταν μιλάμε για τις μεταβατικές διατάξεις και μιλάμε για τον κανονισμό 13 ε, του 2013 θα πρέπει να επαναξεταστούν αυτές οι αρχές. Επίσης, όταν μιλάμε για τη δυνατότητα της χρήσης ε, της ε, εθνικής ε, στήριξης ε, στην παράγραφο 37 ε, του κανονισμό 1037 του 2013 και η τρίτη πρότασή μας αυτό είναι κάτι πρέπει να ληφθεί υπόψη η μεταβατική περίοδος θα πρέπει ενδεχομένως να πάει στο το 2022 να την ε, παρατείνουμε δηλαδή ευχαριστώ ευχαριστώ και τώρα ο Άλβαρο Αμάρο έχει το λόγο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι ο σκιώδης συγητής του ΕΛΚΑ ε, για αυτό τον κανονισμό και ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ βεβαίως με τον συντονιστή μου, τον κύριο Ντόρφμαν, να υπογραμμίσω όμως μια πτυχή που δεν πρέπει να ξεχνάμε. είναι κάτι που αρχίζει να γίνεται σημαντικό για όλους μάλιστα θα έλεγα. Σε επίπεδο μετάβασης, μεταβατική περίοδο, ένας γεωργός χρειάζεται προλευσιμότητα. Κάποιος είπε για ένα έτος μεταβατική περίοδος ε, της προάλλες. Ε, θα πρέπει να δούμε όμως ε, αν έχουμε, τι θα γίνει αν έχουμε ένα χρόνο μεταβατική περίοδο. Εάν στο τέλος του έτους χρειαστεί ε, άλλο ένα έτος, να μην αρχίσουμε από το μηδέν τη συζήτηση. Ας έχουμε λοιπόν ένα έτος με ένα αυτόματο rollover όμως προς ένα δεύτερο έτος. Ιδάλλως ε, ανοίγουμε την πόρτα σε μια πιο μακροσκελή μεταβατική περίοδο. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Ε, δεύτερον, το οικονομικό σκέλος, τον έφερε και ο συνάδελφος. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Δεν θα ήταν δίκαιο, δεν θα ήταν αποδεκτό στη βιβλιοτική αυτή περίοδο, είτε είναι ένα έτος είτε δύο, η υποστήριξη για τους γεωργούς να μειωθεί. Αυτό δεν είναι μετάβαση. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό κάτι τέτοιο λοιπόν. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε Λοιπόν, ότι τα στοιχεία, τα αριθμητικά, θα είναι τα ίδια. Αυτό είναι κάτι που το είπε ο κύριος Ντόρφμαν και το υποστηρίζω και εγώ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τουλάχιστον τα ίδια αριθμητικά στοιχεία με αυτά που προβλέπονται σήμερα. Τα ίδια ποσά. Εάν έχουμε περικοπές στην κοινωνική πολιτική ε, και στο πολιτισμικό πλαίσιο, ε, αυτό θα ήταν λάθος. Δηλαδή, περικοπές στην πολιτική συνοχή γενικά σημαίνει λιγότερη αλληλεγγύη. Θα επηρεαστούν οι πολιτικές μας. Θα έχει αντίκτυπο αυτό. Και θα είναι ακόμα πιο άδικο βέβαια οι γεωργοί να αναλάβουν το βάρος αυτής της μετάβασης μέσω περικοπών. Αν η κοινωνική πολιτική ολοκληρωθεί σήμερα, θα έχουμε μια άλλη κοινωνική πολιτική αύριο. Ωραία. Αλλά δεν πρέπει να το πληρώσουν οι γεωργοί αυτό. Δεν πρέπει αυτοί να υπομισθούν το βάρος της μετάβασης. Ακούσαμε για τι πλέον αποκλεισμένες περιοχές, ε, για την ανάπτυξη τη υπέτρο και αυτά είναι σημαντικά. Και ο δεύτερο πυλώνα. Είναι μια κρίσιμη πτυχή γενικότερα, ένα κρίσιμο, μια κρίσιμη στιγμή για τη γεωγραφική ισορροπία στην Ευρώπη. Το είπα και χθε, το παραλαμβάνω και σήμερα. Εγώ υποστηρίζω 100% την ιδέα αυτή, το σχέδιο από την εκμετάλλευση στο πιάτο. From farm to fork. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι για να φτάσει στο πιάτο χρειαζόμαστε την εκμετάλλευση πρώτα για να φτάσει στο πιάτο του προϊόν. πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε οπωσδήποτε ιδιαίτερα ε, τις πιο μειονεκτικές περιοχές της Ευρώπης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριος Πεκάινεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι σε 45 εβδομάδες Πρέπει να ισχύσει η νομοθεσία για τη μεταβατική περίοδο και να βασίζεται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Αυτό έχει γίνει νομίζω και στο παρελθόν. Ε, πριν από χρόνια νομίζω τα πράγματα αυτά είναι συνηθισμένα μέτρα. Δεύτερον, θέλω να τονίσω ότι δεν θα δεχτούμε περικοπές ε, στην ΚΑΠ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι αγρότες μας είναι η ραχοκοκαλιά της υπαίθρου και να τονίσω πόσο σημαντική είναι η γεωργία για τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Οι αγρότες ε, κρατάνε την ύπεθρο ζωντανή. Τρίτον, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς ιδιαίτερο λόγο άφησε εκτός των προτάσεων της ε, οποιαδήποτε μετραγία εθνική μεταβατική βοήθεια και εθνικά προγράμματα τα οποία είναι κομμάτι του πακέτου βοηθεία στην ΚΑΠ. Παραδείγματο χάρη στη Φιλανδία. Από όταν μπήκαμε το 1995 συνεχίζονταν η εφαρμογή αυτών των μεθόδων και πρέπει να συνεχιστεί και τώρα, ειδικά στην μεταβατική περίοδο. Τώρα, εάν και όταν συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε ε, τους υφιστάμενους κανόνες πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί και η εθνική ενίσχυση και το είπαν και δύο συνάδελφοι ελπίζω να το τονίσει και η Επιτροπή στη γνωμοδότηση ελπίζω να ολοκληρώσουμε γρήγορα έτσι ώστε η Επιτροπή Γεωργίας να προχωρήσει το στόμα τον Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ντανιέλ Μπούντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπωσδήποτε στηρίζω τον κύριο Ντόρφμαν και τους και γιατί οπωσδήποτε ε, χρειάζεται τη στήριξη η γεωργία για να έχει και την δυνατότητα να παρέχει ποιοτικά τρόφιμα για όλους. Συνάδελφοι, τα είδαμε αυτά σε συζήτηση με άλλους συναδέλφους που ίσως να μην γνωρίζουν το τι γίνεται ε, στα θέματα αυτά. Ε, γιατί θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια λογική χρηματοδότηση για την πολιτική γεωργίας και συνοχής. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί χωρίς σταθερή χρηματοδότηση της ΚΑΠ οι τιμές των τροφίμων θα ανέβουν τόσο πολύ ώστε πολλοί κόσμος δεν θα μπορεί να, να φάει. Έχουμε λοιπόν έναν ανεπτυγμένο τομέα γεωργικό που παρέχει ποιοτικά τρόφιμα ε, θα ευτυχώς από εισαγωγές από άλλες χώρες. Χρειαζόμαστε λοιπόν χρηματοδότηση στις ε, απομακρυσμένες περιοχές. Είχα πάει στην προηγούμενη θητεία στις Αζόρες και στην Μαρτινίκα και βεβαίω πράγματι πρέπει να έχουν σταθερή χρηματοδότηση από την Ένωση ταυτόχρονα. Θα ήθελα να τονίσω αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος. Πρέπει να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να δώσουν μεταβατική εθνική στήριξη, γιατί αυτή είναι πόρη που δίνει ο εθνικός περιβολισμός και όχι τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και πρέπει να τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν τη στήριξη. Τέλος, να τονίσω την ανάπτυξη της υπαίθρου. Μιλάμε για τον δεύτερο πυλώνα. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λεφτά από την πολιτική συνοχής για να εξυγχρονίσουμε τις περιοχές της υπαίθρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εάν σκεφτούμε την συνέργεια των κονδυλίων τότε οπωσδήποτε θα έχουμε λεφτά να αναπτύξουμε τις περιοχές αυτές και οπωσδήποτε βεβαίω. πρέπει να υπάρχει μια καλή συνέχεια της χρηματοδότησης για την ΚΑΠ και την πολιτική συνοχή. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μορτανόφσκα έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για μαθηματικές διατάξεις για την υποστήριξη αυτών των δύο ταμείων, αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτή η διάταξη να μας οδηγήσει να, μετα... να παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο μετά το 2020. Είναι σημαντικό αυτό. Η μεταρρύθμιση του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου ε, μπορεί να μην τεθεί σε ισχύ από το Σεπτέμβριο του 2020 ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και η εθνική υποστήριξη και να στον κανονισμό 1037 του 2013. Επίσης χρειάζεται ευελιξία. Το 25% να μπορεί να, μετα... μετακινηθεί, να μεταφερθεί μεταξύ πυλώνων. Οι μεταβατικές διατάξεις πρέπει να μας να δώσουν και τη δυνατότητα ε, χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα κατόφυλλα για την περίοδο 2014-2020. Είναι σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι στο νέο πρόγραμμα, στη νέα προγραμματική περίοδο, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνική συνδρομή. Είναι λοιπόν σημαντικό να εγγυηθούμε αυτή τη δυνατότητα. Σε ό,τι αφορά τα φρούτα και λαχανικά, ε, εδώ ανησυχούμε δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος για τους παραγωγούς. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2021 θα αλλάξουν τα επικοινωνιακά προγράμματα ε, και θα δούμε αν προσαρμόζονται στις νέες αρχές. Και βεβαίως για την Πολωνία είναι τεράστια η αλλαγή. Ε, πάμε ένα έτος πιο εκεί την εξισορρόπηση των επιμέρους πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Πριν δώσω εκ νέου το λόγο στον εισηγητή μας για να κλείσει τη συζήτηση, έχουμε μαζί μας εδώ και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την DG Agri και την DG Regio. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, αν θέλει να παρέμβει ενδεχομένω και να αντιδράσει στα σχόλια που ακούστηκαν. κυρία Κριστίνα Καράσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να πω. Σας ευχαριστώ πολύ ε, που αντιλαμβάνεστε ε, το πόσο επίγει αυτή η πρόταση. 45 εβδομάδες έχουμε. Ε, συζητήθηκαν, συζητήθηκε περιορισμένος αριθμός θεμάτων και αυτό είναι καλό για να προχωρήσουμε διαπραγματεύσεις οι περισσότερε από τι ανησυχίε σα έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση, με τα χρήματα. Ε, για το επόμενο έτο, τα χρήματα για τη μεταβατική δηλαδή περίοδος, περίοδο ε, αντιστοιχεί, αντιστοιχεί το ποσό αυτό ε, σε αυτά που έχουν προληφθεί στο πι, το ίδιο ισχύει για τι πλέον ομακρυσμένε περιοχές. Επίσης κάτι άλλο που άκουσα και συμφωνώ ότι χρειάζεται σταθερότητα, χρειάζεται προλεψιμότητα για τους γεωργούς, όχι μόνο για τους γεωργούς, για όλη την Ήπεθρο. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα επιφελθούν από τα μέτρα αυτά στις διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Αυτό λέμε και εμείς, αυτό προτείνουμε. Συνέχεια, συνέπεια για το 2021 και για μας επίσης ε, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει κάτι γρήγορα για να καλύψουμε τις ανάγκες εντός ενός έτους Οπότε περιορίστε τον αριθμό των ετοιμάτων. Σημειώσαμε βεβαίω ε, κάποια από τα αιτήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι μεταβατικέ ενισχύσει σε καποια κρατημέλη, τη Φιλανδία, τα επιχειρησιακά προγράμματα για τα φρούτα και λαχανικά. Είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε όλα αυτά με τα δύο θεσμικά όργανα για να σα υποστηρίξουμε τεχνικά και διάφορα τον τριλόγου. Ευχαριστώ πολύ για το πόσο γρήγορα εξετάσετε το θέμα αυτό. Είναι απαραίτητο όμω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, δεν ε, χρειάζεται να πω πολλά. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευρεία συμφωνία. Το σημαντικότερο ίσως είναι η διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Έχουμε μια λύση ένα συν ένα που προτείνεται από τους συναδέλφους. Ίσως θα ήταν λογικό να περιοριστούμε δηλαδή στο ένα έτος, αλλά να προβλέψουμε ήδη ότι χρειαστεί άλλο ένα έτος να είναι απλή η παράταση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό, δεν ξέρουμε πότε θα ψηφίσουμε για την ΚΑΠ, αλλά να νομίζω δεν είναι ιδεώδες να ψηφίζουμε μεταβατικό διάστημα δύο χρόνων αλλά καλό είναι να ψηφίσουμε για ένα έτος και άλλο ένα εάν αυτό χρήστη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σημείωσα ότι τελικά όλες οι πολιτικές ομάδες συγκλίνουν ε, όλες δηλαδή ακολουθούν ουσιαστικά τη γραμμή του εισηγητή στην εισαγωγή του. Να θυμίσω ότι η ψηφοφορία προβλέπεται 2 Απριλίου στο Στρασβούργο στην Επιτροπή μας και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι ε, η Δευτέρα 2 Μαρτίου 5 το απόγευμα. Ε, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 8 της ημέρας διάταξης ε, το 7 το αφήνουμε μιας και ο συνάδελφος Λαγουτιγού που ήταν να παρέμβει δεν είναι εδώ ελπίζω να εμφανιστεί αργότερα ε, να περάσουμε λοιπόν στο σημείο 8 της ημέρας διάταξης ε, με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τον Φρεντερίκ Βαλιέ ο οποίος είναι εδώ όπως ξέρω γενικό γραμματέα ε, του CCRE. Ξέρετε ότι το, το Συμβούλιο Κοινοτήτων και Περιφερειών της Ευρώπης είναι η πιο παλαιά, η πιο σημαντική ένωση ε, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη. Είναι η μόνη οργάνωση ε, όπου συμμετέχουν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις από 41 χώρες της Ευρώπης σε όλα τα επίπεδα αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αποχωρεί ησύχω, έτσι. Και η βοηθή παρακαλώ ε, να σταματήσουν να μιλούν να μικρόφωνα. Ε, σας ευχαριστώ. Ναι, ίσως είναι κουραστικό. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στο Φρεντρίκ Βαλιέ Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ μαζί μας και θα ξεκινήσει η συζήτηση στη συνέχεια γιατί έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπατε, το Συμβούλιο Κοινοτήτων και Περιφερειών της Ευρώπης ε, είναι η ομοσπονδία των ε, εθνικών ενώσεων ε, τοπικών περιφερειακών αρχών εκπροσωπούμε συνολικά με τα μέλη μας 130.000 δήμους, πόλεις, περιφέρειες, επαρχίες της Ευρώπης, 100.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δύναμη του δικτύου μας είναι η αντιπροσωπευτικότητα, και εκπροσωπούμε και την Ήπεθρο αλλά και τις μεγάλες πόλεις και βεβαίως ε, έχουμε πρόσβαση και στις εθνικές κυβερνήσεις. Οι δραστηριότητε μας ε, έχουν πέντε θεματικές που αφορούν όλες τις πτυχές ε, της καθημερινότητας, της καθημερινότητας των πολιτών. Η διακυβέρνηση, η δημοκρατία, το περιβάλλον, η ενέργεια, η, συνεργασία, η διεθνή συνεργασία, η πολιτική, η κοινωνική και ταφική συνοχή, οι τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες. Η πρώτη μας αποστολή είναι να είμαστε ένα μέρος ανταλλαγής απόψεων, τεχνο, ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών και τακτικά οργανώνουμε έρευνες και δημοσιεύουμε ε, κείμενα ε, σχετικά ζητήματα. Οι πιο πρόσφατε δημοσιεύσει μα στις ε, Σα φέραμε και κάποιε από αυτέ. Έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, το ευρωπαϊκό εξάμεινο στο τοπικό επίπεδο, η ανάλυση των δομών και ε, αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών στην Ευρώπη. Ε, επίσης ε, έχουμε συμμετέχουμε σε σειρά από project από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή, ή και άλλους εταίρους μεταξύ άλλων το πλαίσιο ε, αναφοράς της βιώσιμης πόλης που είναι ένα συνοδευτικό εργαλείο των περιφερειακών αρχών για τα σχέδια δράση τους για την, περιφερειακή, για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη ιδιαίτερα ε, σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί. Η δεύτερη αποστολή μας είναι να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την, την ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, όταν, αυτή, όταν αυτή έχει αντίκτυπο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό είναι και το νόημα της παρουσίας μας εδώ. Εδώ και πολλά χρόνια ε, από την Επιτροπή Ρέτζη και άλλες επιτροπές ε, συνεργαζόμαστε με όλες τις επιτροπές βεβαίως ε, περιλαμβάνουν τον, την, εδαφική, την εδαφική προσέγγιση. Έχουμε και μια εθνική διάσταση και διεθνή διάσταση μάλλον συμμετέχουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο σε μια αντίστοιχη ένωση. Συνεργαζόμαστε με αυτούς, εκπροσωπούμε τα ευρωπαϊκά εδάφη στα Ηνωμένα Έθνη και στους άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΩΣΑ. Επίσης έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σύμπραξη με την DG DEFCO ε, σε ό,τι αφορά την ε, σύμπραξη μεταξύ πόλεων ε, με τις χώρες με αναπτυξιακές με τις χώρες χώρες. Για μας η περιφερειακή, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι στην καρδιά του ευρωπαϊκού σχεδίου, είναι πολύ σημαντικό αυτό και γι' αυτό είμαστε ε, ιδρυτικό μέλος της ε, ε, Συμμαχίας για τη Συνοχή υπό την αιγίδα της, της, της των Περιφερειών. Είμαστε υπέρ μιας πολιτικής συνοχής που, που ανταποκρίνεται στους στόχους που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά χρειάζεται ένας προπολογισμό ε, που να αντιστοιχεί στο ύψος αυτών των φιλοδοξιών. Έχουμε ζητήσει από του Σαρλ Μισελ ένα προπολογισμό για τη συνοχή αντίστοιχο με το 1 τρίτο του συνολικού προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν ε, υποστηρίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ε, Επιτροπή Ρέτζη στι διαπραγματεύσει για το επόμενο πολιτευτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Θεωρούμε ότι οι τελευταίε προτάσει του Συμβουλίου είναι ανεπαρκεί με βάση τι ανάγκε των ευρωπαϊκών εδαφών. Ε, τα μέλη του CCRE έχουν εκφράσει την άποψή του, η οποία συνοψίζεται σε τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα πρέπει γρήγορα να βρεθεί μια λύση στα πλαίσια του επόμενου ΠΔΠ. Βεβαίως ε, έχουμε καταλάβει ε, ότι θα, συμβεί αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει σε οποιοδήποτε αντίτιμο. Η μείωση του προπολισμού τη πολιτική συνοχή δραστικά, όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο πλέον, αντιβαίνει του φιλόδοξου στόχου τη νέας Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οικολογική μετάβαση, η οποία πρέπει να είναι δίκαιη για τα εδάφη και του ανθρώπου. Ε, το νέο Ταμείο για τη Μετάβαση θα πρέπει να έρθει να συμπληρώσετε τα δυτικά ταμεία και επενδύσεων της Ένωσης. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πολλές χώρες ε, ε, θέλουν να μεταφέρουν 1,5-3 φορές το, το ποσό αυτό από το Φέντερ ή το FSE. Εμείς δεν είμαστε υπέρ αυτού του μέτρου, διότι αυτό οδηγεί σε μείωση των δυνατοτήτων δράση από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Φεντέρ. Ε, η προσθέμενη ε, αξία του νέου ταμείου μας φαίνεται ισχνή, μιας και ήδη τα υπάρχοντα ταμεία μας επιτρέπουν να μειώσουμε τις αποστολές, ε, ε, την ανάπτυξη της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας και άλλα, άλλα σχετικά project. Δεν πρόκειται για νέο προπολογισμό. Βέβαια, μια και τα 7,5 δισεκατομμύρια τα οποία έχουν ανακοινωθεί θα προέλθουν από το υπάρχον τα προπολογισμό για την περιφερειακή ανάπτυξη του, του Ταμείου, δηλαδή του ΦΕΝΤΕΡ. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο για την Δίκαιη Μετάβαση, εμείς θεωρούμε ότι είναι καλό ότι οι στρατηγικές καθορίζονται σε επίπεδο ΝΑΤΣ 3, που είναι το, αυτό που είναι πιο κοντά στους πολίτες και το πλέον κατάλληλο για πολιτικές εδαφικής ανάπτυξης βιώσιμες και ολοκληρωμένες. Το Ταμείο αυτό πρέπει στο μέτρο του δυνατού να πάει προς αυτούς που το χρειάζονται, προς τα εδάφη που το χρειάζονται και θα φροντίσουμε να συμβεί αυτό το CCRE προωθεί μια πολυκεντρική ε, προσέγγιση της περιφερειακής ανάπτυξης. Ε, είμαστε υπέρ επίσης ε, οι περιοχές της Υπέθρου να είναι ένας τόπος δυνατοτήτων, ένας τόπος ευκαιριών και να υπάρχει μια συμπληρωματικότητα με την αστική ανάπτυξη, συνεισφέροντας έτσι αρμονικά ε, στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αστικής Ατζέντα, στην οποία επίσης συμμετέχουμε. Το CCRE συμμετέχει στη συναντήσεις των κρατών μελών για την εδαφική ανάπτυξη και την αστική ανάπτυξη. Συνεισφέρουμε έτσι αυτή τη στιγμή στην ανανέωση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Γερμανικής Προεδρίας στα πλαίσια της νέας χάρτας για τις βιώσιμες πόλεις και τη νέα εδαφική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το CCRE συμμετέχει ε, στις συζητήσεις της ε, Πολιτικής Επιτροπής του ΟΣΑ για την περιφερειακή ανάπτυξη, όπου επίσης εκπροσωπούμε την άποψη των τοπικών και, τοπικών και ε, περιφερειακών αρχών. Αυτά ε, σε την παρουσίασή μου, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Φρεντερίκα. Και τώρα το λόγο έχει η συνάδελφος Νόρα Μεμπάκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτήν την αποσαφήνιση, γιατί χτες συζητούσαμε το ταμείο, μάλλον προσπαθούσαμε να συζητήσουμε για το Ταμείο Δίκαιης Μετάφασης. είναι λοιπόν διαφωτιστικό αυτό το σημείο να ξέρουμε δηλαδή ποιες είναι οι δημόσιες πολιτικές όσον αφορά τη συνοχή. Αυτά τα θέματα είναι εξαιρετικά σημαντικά για τις διάφορες περιφέρειες. Ε, είναι αλήθεια ότι όταν έφτασα, ε, πριν δύο μέρες μόλις προσγειώθηκα σε αυτήν την Επιτροπή, διαπιστώνω ότι ένας τόσο περιοριστικός και μειούμενος προϋπολογισμός, γιατί αυτό κατάλαβα από τη συζήτηση, δείχνει πως δεν είμαστε στο ύψος των περιστάσεων και κυρίως στο ύψος των περιστάσεων της συνδιακυβέρνησης με τις ε, περιφέρειες. Και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης να μην γίνει απλά ένα κόμμα, ταμείο το οποίο δεν θα έχει τους απαραίτητους πόρους ε, και θα ε, πρέπει να χρηματοδοτηθεί από, άλλους, από άλλα κονδύλια. Εμείς θέλουμε να είναι επιπρόσθετο και όχι ε, οπισθοδρομικό. Ευχαριστώ. Συνάδελφος, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. καλημέρα σε όλους. Πραγματικά το εκτιμώ που η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι σημαντική όσον αφορά την συνοχή, γιατί γίνονται απόπειρες να αποδυναμωθεί η συνοχή. Η χώρα μου ανοίγει στα 16 κράτη-μέλη που είναι φίλοι της συνοχής. Πρέπει να δοθεί αυτός ο αγώνας, γιατί η πολιτική συνοχής αναγνωρίζεται από τους πολίτες, είναι πολύ αναγνωρίσιμη και πιστεύουμε πως είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους νέους στόχους. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή σας τη συνεργασία και να τονίσω πως είμαστε πιο κοντά έτσι, στους πολίτες και γι' αυτό και τα όσα μας λέτε είναι πολύ σημαντικά. Να έχω μια ερώτηση. Εχθές συζητήσαμε περί του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και θα ήθελα να έχω τη γνώμη των περιφερειών που εξαρτώνται ας πούμε από τον άνθρακα. Πώς ε, θα βλέπουν τις επενδύσεις σε τεχνολογίες ε, οι οποίες είναι και αυτές μεταβατικές όπως για παράδειγμα το φυσικό αέριο γιατί πολλοί είναι κατά οποιασδήποτε χρηματοδότηση στήριξης σε οποιοδήποτε ορυκτό καύσιμο όπως είναι και το φυσικό αέριο. Εγώ από ό,τι κατάλαβα όμως στόχος είναι ε, να συμβούν οι νέοι στόχοι του περιβάλλοντος, για το περιβάλλον μάλλον, και αυτό θα είναι δύσκολο χωρίς τη χρήση του φυσικού αερίου. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ. Ε, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μια ερώτηση προς τους εκπροσώπους των περιφερειών. Στον τύπο διάβασα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης στη στην Πολωνία είναι η Βαρσοβία και στη Γερμανία το Βερολίνο θέλουν να στήσουν ένα συγκεκριμένο κονδύλι το οποίο θα το θα είναι μέσα στις ε, νέες δημοσιονομικές προοπτικές ένα ταμείο ανάπτυξης ε, που θα επέτρεπε σε αυτήν την ένωση μεγάλων πόλεων αστικών κέντρων δηλαδή αυτές θα έχουν στα χέρια τους την αναπτυξιακή πολιτική στις περιφέρειές τους, δηλαδή τις περιφέρειες που συνδέονται με τις πόλεις αυτές. Έχετε πληροφορίες για αυτό το θέμα και αν ναι μπορείτε να μας τις πείτε. Σας ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ και ένα θερμό καλωσόρισμα στους εκπροσώπους των ε, Δήμων και Περιφερειών. Και εγώ έχω διατελέσει δήμαρχος για 30 χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά πώς λειτουργούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που είναι πραγματικά η καρδιά της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για την Επιτροπή των Περιφερειών και για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων να συμπεριλαμβάνονται στην χάραξη των πολιτικών μας. Ε, αφέρατε διάφορα σημαντικά ζητήματα για το νέο PDP. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν είναι πρόθυμοι φυσικά να, να δεχτούν απευθεία το τι μας προτείνεται και αυτό που έχω υπόψη μου είναι κυρίως οι περικοπές στην χρηματοδότηση που σχετίζονται με τη ζωή των και των περιοχών και των περιοχών της υπαίθρου. Η υπαίθρος είναι αυτή που παρέχει, μάλλον το Ταμείο συνεχή είναι αυτό που δίνει τα περισσότερα χρήματα για τη διατήρηση αυτών των δραστηριοτήτων. Γι' αυτό και πρέπει να οργανωθούμε και να εξασφαλίσουμε την ε, χρηματοδότησή τους. Επίσης είμαι ε, της άποψης πως ε, οι περιφέρειες και οι δήμοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημογραφία της Ευρώπης και στη μετανάστευση. Παρακολουθώ αυτά τα θέματα πολύ εκ του συνεγγύς. Είτε πρόκειται λοιπόν για Ανατολική είτε για Δυτική Ευρώπη. Βλέπουμε τι συμβαίνει. Βλέπω τι συμβαίνει στη Βουλγαρία, στην Κροατία, στη Βαλτική. Και σε όλους αυτούς τους τομείς έχουμε και αντιμετωπίζουμε μετανάστευση βλέπουμε ότι ο κόσμος προσπαθεί να μετακινηθεί στην Δυτική και ε, Ευρώπη όπου υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση και εάν δεν καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτές τις εξελίξεις, αυτό σίγουρα θα επηρεάσει τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κόσμος ε, στη Βουλγαρία θα, θα, ρωτά, κατα, θα ρωτά κατά πόσο αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ε, την ξέρουμε. Εάν συγκρίνουμε ανάμεσα στο 2019 και το 2050, τις προοπτικές του 2050, η ευημερία θα μειωθεί κατά 40% και ο πληθυσμός θα μειωθεί κατά 30%. Οπότε οι πολιτικές που υιοθετούμε τώρα θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στη και προσοχή στις πόλεις, γιατί πιστεύω πως αυτά τα ζητήματα θα μας προκαλέσουν πολλούς πονοκεφάλους στο μέλλον ε, να σκεφτούμε λοιπόν νέες ιδέες, νέες αντιλήψεις που θα συνδυάσουν το χώρο για τους ηλικιωμένου, τη φροντίδα για τους ηλικιωμένου και πάντοτε να έχουμε υπόψη ότι πρέπει να αποκεντρωθεί η απασχόληση σε άλλες περιοχές και να στηρίξουμε και εκείνες τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Δυστυχώς όμως όλα αυτά τα πράγματα τα, ε, δεν τα βλέπουμε στην πράξη. Ε, αντίθετα, οι περισσότερε περικοπέ προτείνονται σε αυτέ τι πολιτικέ. Γι' αυτό και είναι δική μα ευθύνη. Όλοι μα πρέπει να συμμετέχουμε και να ασχοληθούμε. πραγματική ζωή βρίσκεται στι περιοχέ τη υπαίθρου και σε αυτέ πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Πρέπει να πω πως εν γέννη συμφωνώ με τα όσα είπατε και στη συνεδρίαση των συντονιστών ε, θα κοιτάξουμε και θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να βασιστούμε στην υπηρεσία έρευνας και μελετών του Ευρωκοινοβουλίου ώστε να έχουμε στοιχεία όσον αφορά αυτές τις δημογραφικές αναταράξεις τόσο παγκοσμίω όσο και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχουν σημαντικές συνέπειες για την συνοχή και τον τρόπο με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε την ε, ε, συνοχή. Όχι σε μακρο, βραχυπρόθεσμα, αλλά σε έναν ορίζοντα 10-20 ετών. Το 2100 ε, υπολογίζεται ότι θα έχουμε 80 εκατομμύρια λιγότερους Ευρωπαίους αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και ήδη και σήμερα βλέπουμε ε, πάρα πολλούς νέους Ευρωπαίους που, ε, που φεύγουν Έχουμε κινήσεις ε, ανθρώπων, συχνά νέων, που φεύγουν από τη μια χώρα στην άλλη. Πάση περιπτώσει, εσύ τα θύμισες όλα αυτά. Είναι πάντως μια υπόθεση καθοριστική και πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια στην Επιτροπή μας να έχουμε μια, μια πιο μακρόπνοη προοπτική. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον συνάδελφο Μόρι. Arvoisa puheenjohtaja, kun paikalla ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Τώρα που είναι εδώ και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής των Περιφερειών, θα ήθελα να σας πω πως ε, η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής ε, έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στις περιφέρειες ΝΑΤΣ 3. Γιατί αυτές ε, αφορούν πολλούς δήμους. αυτό ακριβώς θα πρέπει και όλοι οι Δήμοι να μπορούν να συμμετέχουν, όχι μόνο οι πόλεις, όλοι οι Δήμοι. Πρέπει να εκπροσωπούνται στον φορέα ο οποίος θα λαμβάνει αποφάσεις για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Εγώ είμαι εκπρόσωπος της μεγαλύτερης πόλης στην περιφερειά μου και λαμβάνω αποφάσεις εδώ και καιρό και παρά το ότι ισχύει αυτό, δεν θεωρώ ότι ε, μόνο εμείς ε, στο κέντρο πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις για τις περιφέρειες. Πρέπει να υπάρχει ένα πραγματικά αντιπροσωπευτικό σώμα. Μέχρι να εκλεγώ λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμουν πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Φιλανδίας. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνει δέκτο στην πολιτική συνοχή να λαμβάνουν μέρος όλοι οι Δήμοι. Σας ευχαριστώ. Θέσαμε τις αρχές της ε, εταιρικότητας, εταιρικής σχέσης ως προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις που είναι υπό εξέλιξη. Είναι μια πολύ ισχυρή γραμμή την οποία υποστηρίζουμε και είναι προφανές ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε οι Δήμοι να συμμετέχουν καλύτερα και περισσότερο μέσα στη διακυβέρνηση. Παντού, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αυτό το αίτημα της ε, εταιρικότητας ε, που δεν τηρείται πάντα. Και βεβαίως πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί τελικά η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση όταν μεταφράζεται σε συγκεκριμένα σχέδια και project ε, προσγειώνονται στις ε, δήμους και ακριβώς οι δήμοι είναι αυτοί που θα πρέπει να ε, περιλαμβάνονται ακριβώς σε όλες τις διαδικασίες καθορισμού και οριστικοποίησης αυτών των ε, ταμείων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλές παρεμβάσεις, πολύ ενδιαφέροντες, ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις. Ίσως όμως πρώτα απ' όλα να άρουμε μια παρεξήγηση. Μιλούσα, άκουσα να γίνεται λόγος για Επιτροπή των Περιφερειών. Δεν είμαστε η Επιτροπή των Περιφερειών. Είμαστε το Συμβούλιο Δήμων και Κοινοτήτων της Ευρώπης και συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά Καμιά φορά ε, τυχαίνει να έχουμε και ελαφρώς διαφορετικές απόψεις, κυρίως όσον αφορά ας πούμε, το σημείο του ΝΑΤΣ 3. Η Επιτροπή Περιφερειών έχει μια θέση νομίζω κάπως διαφορετική από τη δική μας, γιατί ε, ακριβώς προτείνει να στοχευθεί περισσότερο το επίπεδο ΝΑΤΣ 3. Δεν θα ήθελα λοιπόν ε, να υπάρξει σύγχυση. Λοιπόν, καταρχάς όσον αφορά την μετάβαση στις περιφέρειες που ακόμα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την, τον άνθρακα. Είμαστε υπέρ της στήριξης της πρόσβασης στο φυσικό αέριο σε ορισμένε περιφέρειες εφόσον πρόκειται για ε, ένα στάδιο. Θα πρέπει να σας πω ότι μίλησα χτες το βράδυ γιατί είχα κάποια για να, για να μαλέψω ιδέες για τις ερωτήσεις που θα τίθεται σήμερα το πρωί με τον συνάδελφο από την Πολωνία. Ξέρετε πως η Πολωνία καίγεται για αυτό το θέμα και αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται σε ορισμένες περιφέρειες ε, μετακινούνται από τη θέρμανση με τον άνθρακα στη θέρμανση με πετρέλαιο. Ε, όπως καταλαβαίνετε ε, έχουμε ακόμα δουλειά. Ε, μπροστά μας και ε, είναι αλήθεια πως ε, οι Πολωνοί θέλουν να προχωρήσουν, αλλά το φυσικό αέριο εξακολουθεί να είναι μία από τις λύσεις που προτιμώνται στην πολωνική επικράτεια με την επιθυμία να μπορέσουν να αναπτύξουν και ανανεώσιμες πηγές και να επιμείνουν στις πολωνικές αρχές για να μπορέσουν να περάσουν και σε αυτό το επίπεδο. Ε, είναι μια επιπλέον, ε, ένα επιπλέον στάδιο το οποίο θα πρέπει να το στηρίξουμε. Τώρα, για το θέμα την ερώτηση που έθεσε ε, κάποιος για το ταμείο το οποίο θα διαχειρίζονται άμεσα οι περιφέρειες, οι δήμοι μάλλον αν κατάλαβα καλά την πρόταση της Γερμανίας και της Πολωνίας. Εμείς είμαστε προφανώς ε, ε, υπέρ του να διαχειρίζονται τα ταμεία οι δήμοι και παρέρχομαι και στις, στα όσα υπόθηκαν στη συνέχεια. Για το Ταμείο Μετάβασης είναι σαφές ότι δεν επιθυμούμε να είναι ένας τρόπος για να κεντροποιηθεί και πάλι ένα κομμάτι των κονδυλίων που δίνονται κατευθείαν στους Δήμους, δηλαδή ε, να παρθούν χρήματα από την περιφερειακή πολιτική για να δοθούν στα κράτη απευθείας. Εδώ νομίζω πως συμφωνούμε και μπορούμε να έχουμε και τη στήριξη της Επιτροπής Ρέτζη, ώστε να εξασφαλίσουμε πως τα κονδύλια που, πάνε, ε, που προορίζονται για τη μετάβαση θα φτάσουν όντως σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο στο επίπεδο των ε, πιο ενδιαφερόμενων δηλαδή περιφερειών. Το θέμα για την δημογραφική εξέλιξη είναι επίσης ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος. Ε, Βουλευτή μίλησε για την Βουλγαρία, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε και για τι βαλτικέ χώρε για τη Ρουμανία. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο κατά τη γνώμη μα δεν αντιμετωπίζεται και που πρέπει να δουλευτεί. Και εδώ συμφωνώ με τον Πρόεδρο. Ε, αν μπορεί να γίνει μελέτη με τη στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου, φυσικά και συμφωνούμε να συμμετέχουμε, διότι είναι ένα από τα ζητήματα που μας αφορούν και βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Πρέπει να σας πω ότι για την ώρα δεν έχουμε κάνει ιδέα γιατί νούμερα μιλάμε όσον αφορά την μετανάστευση των νέων από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ή ακόμα και πιο μακριά. Και είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Νομίζω σε αυτά θα σταματήσω γιατί δεν θέλω να μονοπολίσω τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή στις εργασίες μας. Τώρα θα περάσουμε στο σημαντικό σημείο της σημερίσιας μας διάταξης γιατί θα συζητήσουμε σε ανταλλαγή απόψε με τον αγαπητό μας συνάδελφο. Μπορείτε να μείνετε αν το θέλετε ε, με τον αγαπητό συνάδελφο Πιέρ Λαρουτουρού που είναι Γενικός Εισηγητής για τον προπολογισμό της Ένωσης για το έτος, οικονομικό έτος 2021. Η φετινή διαδικασία, όπως γνωρίζετε, είναι υποσυζήτηση, υποδιαπραγμάτευση και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2021 μέχρι και 2027 και η Επιτροπή Προϋπολογισμών κάλεσε τις ε, επιμέρους επιτροπές να γνωμοδοτήσουν όσον αφορά το προσανατολισμό και τον προϋπολογισμό του 2020. Ο κ. Λαροτουρού παρουσίασε το σχέδιο έκθεσης του και τους προσανατολισμούς του πριν από δύο μέρες μόλις στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και σήμερα θα μας παρουσιάσει το θέμα ε, εδώ και μετά θα δώσω το λόγο στους εισηγητές, εσκιώδης και τους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ μαζί σας, διότι μιλάμε για την καθημερινότητα εδώ τι γίνεται στις πόλεις μας, στα, στα εδάφη μας, στα χωριά μας και η συζήτηση για τον προπολογισμό είναι βεβαίω σημαντική. Υπάρχει κίνδυνος ο προπολογισμό μας να είναι ανεπαρκής. Είμαι νέος βουλευτής όπως πολλοί από εσά, ε, έξι μήνες ε, θητεία έχω και μου ζήτησαν να είμαι γενικό συζητητή ε, για τον προπολογισμό του 2021. Πριν μπω στι λεπτομέρειε τεχνικέ, νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι το διακύβευμα των πολιτικών είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα πρέπει οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μείνει ενωμένο να θέλουμε να κερδίσουμε τη μάχη για ένα φιλόδοξο προπολογισμό. Ο προπολογισμό του 2020 ε, καταφέραμε εκεί να κερδίσουμε 1,9 δι παραπάνω από αυτά που ζήτησαν οι αρχικοί καλών κυβερνήσεων. Συμμετείχαν πέντε όμω πολιτικέ ομάδε στην συμμαχία αυτή. Ήμασταν ενωμένοι. Φέτο και για το προπολογισμό του 2021 και για το ΠΔΠ θα είναι ακόμα πιο περίπλοκη η μάχη και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι για άλλη μια φορά. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο είναι τι θα γίνει με τα ταμεία συνοχή, πώ θα αποφύγουμε τι περικοπέ. Συνάντησα τον Πέτρο Κώστα στι Βρυξέλλε ε, χθες και συζητούσαμε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πάνε πίσω σημαντικές πολιτικές συνοχής της Ένωσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Οι περισσότεροι, για να είμαι ειλικρινής, θεωρούν ότι το Κοινοβούλιο θα υποχωρήσει. Εγώ, ως Γενικός Εισηγητής, πάω κάθε μήνα στο Βερολίνο. Θα προεδρεύσει ε, η Γερμανία το δεύτερο εξάμεινο. Ε, έχω δει δημοσιογράφους. Όλοι θεωρούν ότι το Κοινοβούλιο, εντάξει, θα γαυγίσει, αλλά στο τέλος θα υποχωρήσει και θα πάρουν ό,τι θέλουν οι αρχικοί καλών κυβερνήσεων. Λοιπόν, εμείς γιατί είμαστε όμως εδώ, ε, απλά για να κάνουμε λίγη φασαρία και μετά τελικά να υποχωρήσουμε ή θα δώσουμε μια πραγματική μάχη. Για να δώσουμε πραγματική μάχη πρέπει να έχουμε επιχειρήματα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει παντού στις Βρυξέλλες και αλλού να βρούμε, να βρούμε περισσότερους πόρους. Ε, νομίζω ότι για, το, για τα ταμεία συνοχής, για την γεωργική πολιτική προφανώς και δεν ε, θέλουμε να υπάρξουν περικοπέ. Ε, εδώ θα συμφωνείτε μαζί μου. Υπάρχουν και νέε προκλήσει όμω. Μια από τι νέε προκλήσει είναι το, το θέμα του κλίματο. Το Green Deal. Ε, το Green Deal είναι σοβαρή υπόθεση ή όχι. Ήμουν στον Παμακό, στο Μαλί πριν από λίγε μέρε, για δύο μέρε. Ε, δεν μπορείτε να φανταστείτε την ξηρασία που υπάρχει στην περιοχή του Σάιλ αυτή τη στιγμή. Είναι μεγαλύτερη εδώ και 1600 χρόνια. Στον Παμακό μα λένε ότι το AIDS μπορεί να, είχε, να έκανε εκατομμύρια, χιλιάδε θύματα μάλλον, αλλά η ξηρασία θα κάνει πολύ περισσότερα. Και αντίθετα από αυτό που πιστεύει κανεί για το κλίμα, παρόλα αυτά που γίνονται στα εδάφη μα, πολλοί κάνουν, πολλά, το ξέρω. Ε, συνάντησα ε, κάποιου επιχειρηματίε το πρωί που κάνουν καινοτομία γύρω από το κλίμα. Κάνουμε πολλά, όμω τα πράγματα χειροτερεύουν. Η... Ε, εδώ βλέπετε τι γίνεται με τι εκπομπέ ε, ε του άνθρακα. Ε, που υπάρχει μια μέτρηση στι ΗΠΑ κάθε εβδομάδα. Αυξάνεται, αυξάνονται εκπομπέ συνεχώ. Και από ό,τι φαίνεται, η, αυτή τη στιγμή η αύξηση είναι τρει φορέ πιο γρήγορη από τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 70. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κανεί να θεωρήσει ότι με αυτά που κάνουμε, αυτά που κάνει η Ευρώπη, οι τοπικέ αρχέ, ε, αλλάζει αυτή η τάση. Όχι, δεν είναι έτσι. Τρει φορέ πιο γρήγορα αυξάνονται οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχει ένα ε, ε, φαύλο κύκλο οι, οι κλιματικές αλλαγές οδηγούν σε πυρκαγιέ ε, στην Πορτογαλία ή στην Αυστραλία. Αυτό παράγει περισσότερο δεξιού του άνθρακα και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη απορρίθμιση. Μα λένε οι κλιματολόγοι ότι μα μένουν λίγα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν η ομιλία τη Ursula von der Leyen έτυχε πολύ θετική αποδοχή όταν είπε ότι το Green Deal είναι προτεραιότητά τη. Το καλό νέο είναι ότι το αυτό το Green Deal, εάν έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μα, θα δημιουργήσει και θέσει απασχόληση. Πολλέ. Λέμε ότι η πραγματική ζωή είναι στην Ήπεθρο. Εγώ είμαι μεγάλο. Επτά χρόνια δίνω μάχη για ένα πραγματικό προπολογισμό για το κλίμα. υπάρχει μια ένωση όλων των χωριών τη της ε, Γαλλία που μα υποστηρίζουν. 10.000 χωριά υποστηρίζουν το σχέδιό μα για τη χρηματοδότηση ενό πραγματικού συμφώνου για το κλίμα. Γιατί λένε τα χωριά μα πεθαίνουν, δεν υπάρχουν θέσει εργασία, υπάρχει απερίμωση, υπάρχει αστιφιλία, υπάρχουν τα κλιματικά προβλήματα. Αν είχαμε τα οικονομικά μέσα για τη μόνωση των, ε, των σπιτιών, για ε, την ε, τηλεεργασία, για μέσα μεταφορά θα μπορούσε να ανασγονεθούν τα χωριά μα. Ζητούμε λοιπόν πραγματικό προβολισμό για το κλίμα. Θα μπορούσε αυτό να δημιουργήσει 5 εκατομμύρια θέσει εργασία στα εδάφη μα, όχι μόνο στι μεγάλε πόλει, αλλά και στι μικρέ πόλει, στι κομοπόλει, στα χωριά που αυτή τη στιγμή πεθαίνουν. Υπάρχει ένα θέμα ισότητα μεταξύ των εδαφών, αλλά και εντό τη κάθε χώρα Υπάρχουν περιοχέ ολόκληρε που πεθαίνουν αυτή τη στιγμή και με μαζικέ επενδύσει στο κλίμα μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση. Μπορούμε επίση να βελτιώσουμε το, την αγοραστική δύναμη. Ε, στην Κρενόμπιλ κάποιο μου έλεγε πρόσφατα ότι ε, σαν το κτίριό μου, είναι πολύ πιο άνετο τώρα για την οικογένειά μου, ζεσταίνομαι λιγότερο το χειμώνα, ε, κρυώνω λιγότερο το καλοκαίρι και κερδίζω και χρήματα στι δαπάνε μου. Αυτό δεν το λέει ένα οικονομολόγο, το λέει ένα απλό άνθρωπο. Κερδίζω κάθε χρόνο 800 ευρώ στι δαπάνε τι ενεργειακέ. Αν είχαμε λοιπόν ένα πραγματικό Green Deal, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε θέσει εργασία σε όλο το έδαφο μα, να επαναζωογονοποιηθούν οι περιοχέ μα και η αγοραστική δύναμη τη κάθε οικογένεια να βελτιωθεί. Το θέμα είναι πώ θα το χρηματοδοτήσουμε το Green Deal, γιατί ο προπολογισμό μα προτείνει αυτή τη στιγμή ο όχι μόνο δεν υπάρχει ένα δι παραπάνω για το κλίμα, υπάρχει μείωση ε, με περικοπέ. Μα ζητούν να κάνουμε περικοπέ στο Ταμείο Συνοχή, στην έρευνα, στον πολιτισμό τη Γεωργία. Είπαμε ότι είναι απαράδεκτο εμεί βέβαια σε όλε τι ομάδε μα. Συνάντησα λοιπόν τον κύριο Κώστα που όπω ξέρετε ε, οργάνωσε μια συνάντηση 17 χρόνων στη Λισαβόνα. Ε, δεν πρέπει να, έχουμε, να επιλέξουμε μεταξύ των Ταμείων Συνοχή και τη δράση για το κλίμα. Πρέπει να βρούμε μέσα ε, έτσι ώστε να διατηρήσουμε το, το Ταμείο Συνοχή και να έχουμε μια φιλόδοξη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το ζήτημα είναι, υπάρχει πολιτική βούληση πέρα από τα λόγια όταν η Ursula von der Leyen κάνει αυτήν την πολύ ωραία ομιλία, την οποία εγώ χειροκρότησα ε, και αναφέρεται στον Κέννεντι, ότι αποφασίσαμε να πάμε στο, στο φεγγάρι. Εντάξει, το είπε ο Κέννεντι, αλλά δεν τα είπε μόνο. Μετά έβαλε και μέσα. Ο προπολογισμό τη NASA πολλαπλασιάστηκε επί 15 τότε. Βεβαίω τραβούσαν τα μαγιά του συλλογιστέ τότε, αλλά σε 4 χρόνια ο προπολογισμό τη NASA πολλαπλασιάστηκε επί 15. Μιλάμε λοιπόν για ένα Green Deal τώρα. New Deal, όπω ο Ρούσβελτ. Βεβαίω, πολιτική αποτελεσματικότητα. Σε τρει μήνε 15 μεταρρυθμίσει τότε, μεταρρυθμίσεις τότε ο Ρούσβελτ. Πραγματικά αλλάζει τα πράγματα. Την ίδια μέρα ε, ψηφίζονται από τα, τα δύο νομοθετικά όργανα οι μεταρρυθμίσει και πολλαπλασιάζεται, τριπλασιάζεται ο προπολογισμό. Και εδώ τώρα μιλάμε για 1,074, 1,078, έτσι. Ο Ρούσβελτ μπορεί να είναι ηλικιωμένο, μπορεί να είναι παράλληλο, αλλά τριπλασιάζει τον προπολογισμό φορολογεί του μετόχου, φορολογεί του πλούσιου, δημιουργεί θέσει εργασία στις πόλεις, στην ύπεθρο για να προστατεύσει τα δάση, για να δώσει αξιοπρέπεια σε όλου του ανθρώπου που ήταν άνεργοι. Ο Κέννη ήταν τρελό, ο Ρούσβελ ήταν τρελό που τα έκανε αυτά. Όχι. Είχαν μια φιλοδοξία και αυτή η φιλοδοξία ακολουθήθηκε από συγκεκριμένα μέσα οικονομικά. Εμεί είμαστε το Κοινοβούλιο, είμαστε η Φωνή των Πολιτών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αρχοί κυβερνήσεων μπορεί να κάνουν πολύ ωραίου λόγου, αλλά δεν ακολουθούν μετά τα λόγια του με συγκεκριμένα μέσα και πρέπει να του πιέσουμε για να το κάνουμε. Αν θέλουμε να πετύχει το Green Deal είναι τεράστια προσπάθεια. Εάν θέλουμε να διαιρέσουμε δύο το διεξίδιο του άνθρακα. Εγώ ήμουν στην ΕΟΚΕ την πρώτη προάλλε και έλεγε ένα εκπρόσωπο επιχειρήσεων ότι δεν περίμενε ε, να ακούσει μια, ένα τόσο συγκεκριμένη δημοκρατική ε, ομιλία. Πρέπει να μονώσουμε τα μισά σπίτια στι πόλεις μα, να κάνουμε, ε, δημιουργήσουμε μέσα μεταφοράς ε, εκεί όπου δεν υπάρχουν, να βοηθήσουμε τους πολίτες στα σχέδιά τους με επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δείτε το έγγραφο 14η Ιανουαρίου, είναι πολύ ενδιαφέρον το έγγραφο αυτό. Διότι Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια λέει ότι εάν θέλουμε να πετύχουμε το Green Deal, θα χρειαστούμε 300 με 600 δι κάθε χρόνο. Το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό. Και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει για την ώρα τα μόνα χρήματα που έχουμε είναι 7 δις από το Ταμείο Δίκες ε, ε, Μετάβασης. Και δεν ξέρω καν αν υπάρχουν όταν διαβάζει κανείς τα που λέει ο Δεν ξέρουμε αν υπάρχει φρέσκο χρήμα δηλαδή. Πού θα βρεθούν τα ποσά αυτά. Διότι αυτά που προτείνονται αυτή τη στιγμή είναι γελία ποσά. Θα πρέπει να καινοτομήσουμε. Ε, Ιδάλω, ε, αυτό που έχουμε μπροστά μα είναι πραγματικά ψίχουλα. Μιλούσα με ένα Πολωνό βουλευτή τη στιγμη ειναι γελια ποσα θα πρεπει να καινοτομησουμε ε ιδαλω αυτο που εχουμε μπροστα μα ειναι πραγματικα ψιχουλα μιλουσα με ενα πολωνο βουλευτη τη προάλλης, μου έλεγε: Έχουμε 30 ορυχεία στην Πολωνία. Για να κλείσουμε ένα ορυχείο χωρί κοινωνική καταστροφή, χρειαζόμαστε 500 εκατομμύρια. Πώ θα χρηματοδοτήσουμε την προσπάθεια αυτή. Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Πολωνία, αφορά και τη Γερμανία, αλλά και την Ισπανία, τη Αστούρια. Υπάρχουν ορυχεία. Και δεν είναι μόνο τα ορυχεία, είναι το σύνολο τη οικονομία που πρέπει να αλλάξει. Ε, μια ολόκληρη ήπειρο. Πού λοιπόν θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε, πώ θα έχουμε αυτό το μετριασμό. Δεν υπάρχει μαγική λύση. Πρέπει να έχουμε ένα όσο γίνεται πιο σημαντικό προπολογισμό και η Επιτροπή Προπολογισμού έχει ξεκινήσει ήδη ακροάσει έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να προτείνει νέε ιδέε. Τρει προτάσει. Πρώτον, μια μάχη για μια πραγματική τράπεζα για το κλίμα. Μα είπαν και βεβαίω χειροκροτήσαμε ότι θα υπάρξει μια τράπεζα για το κλίμα που θα χρηματοδοτεί τι τοπικέ αρχέ για τη μόνωση, τι μεταφορέ. Όμω για την ώρα αυτή η τράπεζα είναι ισχνή. 16 δι. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διπλασιάσει τα δάνειά τη. Ωραία. Για το κλίμα. Πολύ ωραία. 16 δις όμως είναι, κάθε χρόνο παραπάνω. Ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ποτέ δεν είχε τόση ρευστότητα. 16 δις μόλις, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο έχει 1.200 δις με το quantitative easing. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, παρακαλώ όμως να ολοκληρώνετε διότι έχουμε μια πολύ φορτωμένη μέρη διάταξη. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ρευστότητα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάει στην κερδοσκοπία. Αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε αλλού. Χρειαζόμαστε επίση ιδίου πόρου. Πάω λίγο πιο γρήγορα. Έχω λιγότερο χρόνο από ό,τι περίμενα. Οι ε, ίδιοι πόροι λοιπόν. Τα περισσότερα κράτη-μέλη, βεβαίω είχαμε το Brexit, ε, αλλά, αλλά τι γίνεται. Οι 27 χώρε που μένουν είναι 27 Θάτσερ που λένε Εγώ δεν βάζω άλλα χρήματα. Ε, θα πρέπει κάτι να γίνει για του δύο σπόρου πιο πολύ σημαντικό προπολογισμό δηλαδή για το κλίμα, για το Ταμείο Συνοχή, χωρί να ζητούμε όμω χρήματα για τα κράτη-μέλη. Πώ θα γίνει αυτό, Μια φορολόγηση τη κυροζήνη. Όχι να απαγορεύσουμε το αεροπλάνο, αλλά σε όλε τι χώρε ε, υπάρχει φορολόγηση στα καύσιμα. Γιατί να μην έχουμε ε, ένα φόρο στην κυροζήνη. Ε, είναι μια πλαστικό φόρο, αφορά όλη την Ευρώπη και βεβαίω αντιμετωπίζει και τον φορολογικό ανταγωνισμό και τη φοροδιαφυγή. 45% ήταν ο φόρο ε, στα κέρδη και τώρα είμαστε στο 19%. Όταν ήμουν εγώ παιδί ήταν 45%, ενώ τα κέρδη αυξάνονται. Ε, Βεβαίω, αυτό σημαίνει ότι πάνε καλά επιχειρήσει, αλλά το θέμα είναι πού πάνε αυτά τα κέρδη. Τα μοιράζονται με του ε, εργαζομένου, ε, θα υπάρξουν επενδύσει ή πάνε στου μετόχου. Ε, και οι μέτοχοι επενδύουν μετά ή πάνε στι χρηματαγορέ. Και ακόμα και το Δούνο του μα λέει σήμερα ότι το μέρο των κερδών που δεν επανεπενδύεται και που πάει στι χρηματαγορέ είναι ένα τεράστιο μακροοικονομικό πρόβλημα. Είναι εντυπωσιακό. Βλέπουμε ότι ε, αυτή τη στιγμή τα μερίσματα αυξάνονται και οι φόροι μειώνονται. Ο Μάριο Μόντι στην έκθεσή του, και το είχε θέσει και ο Ζάκ Ντελόρ αυτό, είναι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την, ε, το φορολογικό ανταγωνισμό. Να έχουμε ευρωπαϊκή φορολογία χωρί να πλήττονται οι φτωχέ οικογένειε, οι μικρέ επιχειρήσει, να μην φορολογήσουμε τι μικρέ επιχειρήσει. Βλέπετε εδώ στην Ευρώπη έχουμε πέσει το 19% στη φορολόγηση. Στι ΗΠΑ, στο Ρούσβελτ, στον Τραμπ, είχαμε 38%. Τελειώνω, Πρόεδρε. Ε, αν έχουμε ένα πραγματικό προπολογισμό, σημαίνει ότι κάθε οικογένεια, το κάθε χωριό θα έχει ευρωπαϊκέ ενισχύσει και δεν θα πρέπει να έχουμε περικοπέ στο Ταμείο Συνοχή. Θα έχουμε νέα εργαλεία ώστε κάθε οικογένεια, κάθε χωριό να έχει ενίσχυση για να δημιουργεί θέσει απασχόληση και να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Αυτά, Πρόεδρε, πρέπει να δώσουμε μια μάχη. Επιμένω. Όλοι νομίζουν ότι το Κοινοβούλιο θα υποχωρήσει. Θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να έχουμε συγκεκριμένε λύσει. Νόμιζα ότι είχα περισσότερο χρόνο, Πρόεδρε, και συγγνώμη πρέπει να μείνουμε ενωμένοι για να μετωπίσουμε, για να υπηρεστούμε τι λύσει αυτέ, να έχουμε ένα πιο φιλόδοξο προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε, να προχωρήσουμε σε ακροάσεις ε, να οργανώσουμε ακροάσει για το νέο πράσινο σύμφωνο, αλλά η σημερινή μας δουλειά είναι πολύ πιο ταπεινή, γιατί πρέπει να εξετάσουμε τη δική σας ε, γνωμοδότηση, τη δική μας γνωμοδότηση για τον προπολογισμό 2021. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, αλλά φοβούμε πως ο προπολογισμό του 2021 είναι πολύ περιορισμένο για να δούμε και όλου αυτού του προσανατολισμούς.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 Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Προπολογισμών που είναι παρόν σήμερα στην Επιτροπή ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ για αυτή σας την εισήγηση, την ευρύτατη που μας εξήγησε καλά τι είναι απαραίτητο. Το 2021 είναι περίπλοκη χρονιά, μια τελευταία χρονιά των παλιών δημοσιονομικών προοπτικών και η πρώτη των νέων. Ε, έχουμε τις πιστώσεις, τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων, τις αναλήψεις ε, δεσμεύσεων κτλ. Ε, πολύ ιδιαίτερη ε, χρονιά και επιπλέον οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα πρέπει να μιλήσουν ε, για τα επόμενα 7 χρόνια μέχρι το 2027. Εξαιρετικά σημαντική φάση γιατί πρέπει να εγγυηθούμε νέα κονδύλια και ένα καλό προπολογισμό για τη συνέχεια έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε ως κρατημέλη στις νέες προκλήσεις. Ένας προπολογισμό που θα βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πολιτική συνοχή που έχει συγκεκριμένου στόχου, εγγυάται την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, δημιουργεί θέσει απασχόληση, επιτρέπει τι συναλλαγέ σε όλες τις περιφέρειες και αυτά όσα είπε ο Πρόεδρος με παρηγορούν ότι θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι ώστε το Ταμείο Συνοχής να μην αμφισβητηθεί. Βλέπουμε το τι συμβαίνει, μιλάμε για δίκαιη μετάβαση, για 7 δις. Είναι πολλά λεφτά, είναι κονδύλια τα οποία παίρνουμε από κάποια προγράμματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την πολιτική Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ξεχνάμε. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ε, δεν μπορεί να είναι ένα ανώτατο όριο για κάθε χώρα. Δεν μπορούμε να περιορίζουμε τα κράτη-μέλη μόνο και μόνο επειδή έφτασαν στην απορρόφηση του μέγιστου ποσού. Θα δώσω λοιπόν τώρα στο, το λόγο στους συναδέλφους γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο περίπλοκη και πιστεύω πως μαζί θα αγωνιστούμε έτσι ώστε ο προπολογισμό του 20 να είναι καλός για μας και κυρίως για την πολιτική ε, ανάπτυξη, την περιφερειακή πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα ο σκιώδης ε, του ΕΛΚ Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο, όχι. Οπότε θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ερικ Μπερξίστ για ε, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Σας ευχαριστώ πολύ, Πιέρ. Ευχαριστώ και τους σκιώδης εισηγητές. Όπως ακούσαμε είναι περίπλοκη κατάσταση με τον προπολογισμό ενός έτους και το νέο πι που ξεκινάει. Ο Φρανς Τίμερμανς ε, είχε πει τις προάλλες ότι το θέμα δεν είναι να σώσουμε τον πλανήτη. Το θέμα είναι να σώσουμε την ανθρωπότητα. Ο πλανήτης θα επιζήσει ούτως ή άλλως. Ε, χαίρομαι λοιπόν που λέτε ότι το θέμα είναι η προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έλεγα ότι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία στο Green Deal είναι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Και θα ήθελα να τονίσω και την κοινωνική διάσταση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης γιατί είναι δύσκολο να δημιουργηθούν νέες δουλειές στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες ε, και τα λοιπά, Αλλά είναι σχετικά απλό να ε, επανεκπαιδευτεί ο κόσμος ε, για να γίνει η ζωή του ευκολότερη όταν θα κάνουμε αυτή την απαραίτητη μετάβαση. Το ένα είναι αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω. Το άλλο βεβαίω είναι ότι έχουμε τα μέσα Και το ερώτημα είναι, έχουμε αρκετά λεφτά στα ταμεία συνοχής, θα έχουμε νέα κονδύλια στο ταμείο δίκαιη μετάβαση ή θα χρηματοδοτηθεί με περικοπές από την συνοχή. Γιατί τότε νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Κάτι άλλο σημαντικό βεβαίως ε, είναι τα ορυκτά καύσιμα που έχουν και μια γεωγραφική διάσταση όταν προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να τα αντικαταστήσουμε με άλλα καύσιμα φιλικά προς το κλίμα και να δούμε βέβαιως πώς θα επηρεαστεί η γεωγραφία με έναν φόρο κυροζήνης και τα λοιπά. Θέλω να το δούμε αυτό. Τέλος. στο το εξή αν επιτύχουμε να σώσουμε την ανθρωπότητα δηλαδή χρειαζόμαστε τα κατάλληλα κονδύλια και αυτά που μας λέει τώρα η Προεδρία του Συμβουλίου δεν αρκούν πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και αυτό το οποίο ακούστηκε επίσης ήδη οι πόροι ευχαριστώ κύριε Πεκάινεν για την ομάδα Ρινιού. Ναι, στα φιλανδικά θα μιλήσω. Κοιτάξτε, είναι μια ιδιαίτερη χρονιά η ΔΕΛΤΑΠΗ ολοκληρώνεται, θα έχουμε νέε πραγματικότητες και πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα τώρα. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι το θεμελιώδες καθήκον που έχει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής Υπάρχουν δηλαδή οι δυνατότητες να κλείσει το χάσμα μεταξύ των περιφερειών. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχουμε μια κατάσταση όπου οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών έχουν μειωθεί, αλλά οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών έχουν αυξηθεί. Ελπίζω η διαδικασία αυτή ε, σημαίνει ότι η Επιτροπή μας και η Επιτροπή Προπολογισμών θα προσπαθήσει να μειώσει τις διαφορές ε, μεταξύ των περιφερειών εντός των κρατών μελών. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε έναν προπολογισμό που θα συνδέεται στενά με τον ορίζοντα και την καινοτομία. Με μια σωστή πολιτική καινοτομίας μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα κοινοτομία που θα προωθήσει μετά την πρόοδο της Ευρώπης. Ένα άλλο θέμα σχετίζεται με την πολύτιμη δουλειά που είχε ξεκινήσει ε, κατόπιν πρωτοβουλία του Ζαν Κλοντ στην προηγούμενη επιτροπή. Μια έμφαση δηλαδή στην ρακτική Θα πρέπει λοιπόν αυτό να φαίνεται σε μέτρα που δημιουργούν σταθερότητα και να περιληφθούν στην πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ η ομάδα ID. Δεν μα γνωστοποίησε τους ε, σκιώδει. Ποιο ε, θα ήθελε να πάρει το λόγο τώρα ε, που γυρίζει. Μάλιστα, ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Το πραγματικό ζήτημα είναι ότι υποσχέθηκαν ε, ε, ένα κονδύλι για να χρηματοδοτηθεί το πράσινο σύμφωνο, αλλά αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Ε, και μετά μιλάμε για την πολιτική συνοχής, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί και βλέπουμε ότι γίνεται λίγο ε, ό,τι να είναι, γιατί στην αρχή ακούστηκαν διάφορα ωραία λόγια από πλευράς της Επιτροπής, όλοι που χειροκροτήσαμε. Ε, είχαμε και μια δεύτερη σκέψη, ήμασταν λίγο επιφυλακτικοί, αλλά καθώς προχωράμε δυσκολίες υπάρχουν και είναι αντικειμενικές. Χρήματα δεν υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχουν. Για το θέμα της κυροζήνης να σας πω ε, ότι και αυτοί οι φόροι θα βαρύνουν τους καταναλωτές, τους πολίτες, τους χρήστες, αυτούς που ήδη έχουν γονατίσει από τους υπερβολικούς φόρους που πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πως ο υπερβολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δίνει ας πούμε διάφορα δισεκατομμύρια για τι πολιτικέ τις πολιτικές ε, και γειτονία, ενώ θα έπρεπε να είναι αυτά πόροι που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ε, διαφορετικά. Με όλη τη σεβασμό κάνω αυτό, την πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα για μένα δεν ξεκινάμε με το δεξί. Ε, προσπαθούμε να κάνουμε όπως το παιχνίδι με τον παπά και να μετακινούμε λεφτά από το ένα κονδύλιο στο άλλο. Για να δούμε λοιπόν από πού θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφήνεια για τίποτα. Περιμένουμε να δούμε. Ευχαριστώ πολύ, Μόνικα Βανά είναι αλήπη. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον Δημήτρη Παπαδημούλη, ε, εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Πρόεδρε, σήμερα σε λίγες ώρες συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής και η πρόταση του Προέδρου Σαρ Μισελ για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από ευρωπαϊκή τσιγκουνιά των κυβερνήσεων. Διότι προτείνουν έναν προϋπολογισμό που είναι αδύνατο να χρηματοδοτήσει αυτά που οι ίδιες οι κυβερνήσεις έχουν υποσχεθεί στους πολίτες τους, που είναι αδύνατο να χρηματοδοτήσει αυτά που η ίδια η Κομισιόν και η κυρία Φόντερ Λάιεν υποσχέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο για τα επόμενα πέντε χρόνια για να πάρει ψήφο εμπιστοσύνη. Και μέσα σε αυτή την ευρωτσιγκουνιά του Συμβουλίου πρωτοστατούν οι πιο πλούσιες και οι πιο ισχυρές χώρες οι οποίες ισχυρίζονται ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερα λεφτά και αυτό είναι ψέμα. Και αυτό είναι εξαπάτηση των πολιτών. Και εδώ δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας. Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή κύριο Λαρουτηρού ότι πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλες οι πολιτικές ομάδες να μείνουν ενωμένες και να διεκδικήσουν τον προϋπολογισμό και για το 2021 του 1,3% και για όλη την περίοδο. Γιατί πολύ απλά για να γίνουν πράξη αυτά που έχουν θέσει ως στόχο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα χρήματα που έχουμε υπολογίσει ε, με την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι είμαστε ενωμένοι και η πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου έχει υιοθετηθεί με πάνω από 90% στην Ολομέλεια. Αλλά πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την πρόταση και να στείλουμε σήμερα ένα μήνυμα στις κυβερνήσεις ότι αν λογαριάζουν ότι θα εκβιάσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το επιχείρημα των καθυστερήσεων και του χρόνου, είναι γελασμένοι. Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο κύριος Σασόλη, είπε καθαρά «Μας χωρίζουν με την πρόταση του Συμβουλίου 230 δισεκατομμύρια για τα επόμενα 7 χρόνια. Για να συναντηθούμε πρέπει να κάνουν βήματα προς την πλευρά μας και το κλειδί εδώ είναι να μείνουμε ενωμένοι. Και για να μείνουμε ενωμένοι πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα πολύ σαφές, καμία περικοπή στις πολιτικές συνοχής, καμία περικοπή στην κοινή αγροτική πολιτική, πραγματική ενίσχυση όπως έκανε ο Ρούσβελτ για το Green Deal, αλλιώς είναι κοροϊδία, και με πραγματικά χρήματα και αύξηση των ιδίων πόρων να χρηματοδοτήσουμε τις καινούριε ανάγκες που η ίδια η Κομισιόν και το Συμβούλιο ζητούν να υλοποιηθούν. Με αυτό το πνεύμα θα καταθέσουμε τροπολογίες στην γνωμοδότηση της περιφερειακής πολιτικής ε, και ελπίζω ότι η σημερινή ενότητα θα διαρκέσει και δεν θα έχουμε ομάδες πολιτικές που στην πορεία θα αποστούν και θα εγκαταλείψουν αυτή την ενότητα ή θα την υπονομεύσουν. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Νομίζω ότι υπόθηκαν όλα. Δεν υπάρχουν δύο μήνυματα, υπάρχει ένα. Το οποίο το συνόψισε πολύ καλά και ο κύριος Παπαδημούλης μόλις τώρα, αλλά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η διαπραγματευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής ε, ε, μάλλον της Επιτροπής Προπολογισμού εάν η του Τσάρλ Μισελ δεν αλλάξει εάν δεν μετακινηθεί εάν δεν προσεγγίσει τη θέση του Κοινοβουλίου τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενωμένα και αποφασισμένα δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί με αυτή την πρόταση είμαστε βεβαίω διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να συζητάμε και να διαπραγματευόμαστε. Αλλά αυτό που διακυβεύεται σήμερα και αύριο είναι κρίσιμο για το μέλλον της Ευρώπης. Θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα εδάφη μας τα επόμενα δέκα χρόνια. Στην περιφερειακή πολιτική μας. Σας δίνω το λόγο για δύο λεπτά, διότι μετά θα είμαι υποχρεωμένος να σας διακόψω διότι συνεδριάζουν και συντονιστέ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σα, συμφωνούμε επί τη ουσία. Ε, κρίση για την κρίση πληρωμών, ακούστε, είναι πιο μικρή, μικρός κίνδυνος από πριν από 7 χρόνια. Ζητήσαμε βεβαίω 184,7 δις ε, για το επόμενο έτος ε, για τις πληρωμές. Πέρασαν από τον ίσιν 2 στον ίσιν 3. Τα, οι πληρωμές δηλαδή είναι πιο ε, σε πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Λένε ότι είναι λιγότερο ο κίνδυνο, αλλά βεβαίω έχουμε ζητήσει τα χρήματα αυτά για να μην υπάρξει κρίση. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση, ρωτάνε όλοι αν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Η απάντηση είναι όχι. Τρει φορέ όχι. Ήρθαν 300 εργαζόμενοι από την τομέα του Χάλιβα, από τη Γερμανία, στι Βρυξέλλε πριν από λίγο καιρό. Μα είπαν θέλουμε να παράγουμε ε, Χάλιβα με λιγότερο δεξιό του άνθρακα. Περπάτησαν για να έρθουν ω εδώ, με στη βροχή και μας, για το φάκελο αυτό, για το χάλιβα, μας είπαν χρειάζονται 2 δις. Η Πολωνία χρειάζεται 30 δις. Ε, η απάντηση λοιπόν προφανώς και είναι όχι. Τα 7 δις, αν αυτό το φρέσκο χρήμα είναι 7 δις για 7 χρόνια, ένα δις το χρόνο δηλαδή, είναι γελίο το ποσό αυτό. Και δεν είναι καν σίγουρο ότι θα τα έχουμε. Το Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να το πει αυτό, ότι είναι γελίο αυτό που προτείνεται. Και το Κοινοβούλιο, όπως είπε και η Γιουνούς, πρέπει να μπορεί να πει όχι το Αγγλικό Κοινοβούλιο ε, έγινε πραγματικό κοινοβούλιο όταν μια μέρα είπαν όχι θέλουμε να ελέγξουμε ίδιους πόρους. Οι Λόρδοι τότε βέβαια ε, στο όνομα του κοινού καλού μπλόκαραν τον προπολογισμό. Είπαν εμείς είμαστε το κοινοβούλιο θέλουμε άλλους πόρους. Είχαμε κρίση έξι μήνες, ένα χρόνο και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε πραγματικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο ρόλο του Κοινοβουλίου, είναι και το θέμα τη συνοχή των εδαφών, είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματο, δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη, έτσι. Α πάρουμε έξι μήνε παραπάνω για να βρεθούν νέοι πόροι. Με ε, ε, είδα τι έλεγε η Κομισιόν πριν από πέντε χρόνια για την φορολόγηση των ε, συναλλαγών των χρηματιστηριακών. Όταν αγοράζω εγώ τυρί, γάλα, σούπερ μάρκετ, πληρώνω ΦΠΑ. Αν βάλουμε λοιπόν ένα φόρο στι χρηματιστηριακέ συναλλαγέ 0,1%. 0,1% μόλι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι αυτό γίνεται σε δύο χρόνια και θα μας φέρει 60 δις το χρόνο. 60 δις, το ξαναλέω. Φόρο 0,1%. Μιλάμε για νέους πόρους, έτσι, χωρίς να αγγίξουμε τους πιο φτωχούς, χωρίς να αγγίξουμε τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. 0,1%. Όλοι πληρώνουμε ΦΠΑ. Όλοι πληρώνουμε, φορο, για το καύσιμα. 0,1 λοιπόν στις χρηματικές συναλλαγές. δεν θα σκοτώσει αυτό το χρηματιστήριο, δεν θα τα πνίξει. Η Κομισιόν λέει ότι γίνεται αυτό σε δύο χρόνια και θα μα φέρει 60 δι. Ε, ε, το φόρο πάνω στα κέρδη 20 χρόνια το λέμε χωρίς να κουμπάμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεκάδες δισεκατομμύρια θα μπορούσαμε να έχουμε σε δύο χρόνια γίνεται δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε το κοινοβούλιο τα κράτη-μέλη από ό,τι φαίνεται μάλλον τα κράτη-μέλη δεν μπορούν ε, να, να, να ανανεωθούν δεν μπορούν να καινοτομήσουν ενώ στον ιδιωτικό τομέα το λέμε συνεχώ. Ε, και εδώ μα προτείνουν ψίχουλα συγγνώμη αμακρηγόρησα. Ε, ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μακροπρόθεσμα από τον Ιούνιο και βεβαίω θα μπούμε στα πιο συγκεκριμένα. Ε, να πούμε ότι το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο, θέλουμε περισσότερα, θέλουμε νέου πόρου. Και βεβαίω και τα χρήματα από τι Ευρωπαϊκέ Κεντρικέ Τράπεζε να, να χρησιμεύσουν το κοινό καλό. Να υπάρξει μια ρύθμιση. Όταν ο, ο, ο, ο Μπαράκ Ομπάμα κάνει τον νόμο ΦΑΤΚΑ, πλέον είναι ε, όλε οι τράπεζε διαφανεί στι ΗΠΑ. Λοιπόν, χρειαζόμαστε κανόνε έτσι ώστε το σύνολο του συστήματο του χρηματοπιστωτικού να λειτουργεί υπέρ του κοινού καλού. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας ε, στο έργο μας. Ε, να ευχαριστήσω και την εισηγήτριά μας, την κυρία Μουσκάνοβα, ε, για το δικό της έργο, για την προπαρασκευή της έκθεσής της. Ολοκληρώνεται αυτή η συνάντηση της Επιτροπής μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στις εργασίες μας από χθες. Ευχαριστώ επίσης ε, όλους όσους ε, δεν αφορά η συντονιστών που θα ξεκινήσει τώρα. Παρακαλώ να αποχωρήσετε γρήγορα και ησύχως. Ευχαριστώ.